Kérem Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι θα προεδρεύσω στα Ουγγρικά. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης που είναι δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις κοινέ επιχειρήσεις απομάκρυσης παράνομων μεταναστών από κράτη-μέλη προς το Αφγανιστάν και άλλες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υπουργό Τομπίας Μπίλστρομ εκ μέρους του Συμβουλίου. Uh, äh, äh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να συζητήσω μαζί σας αυτά τα σημαντικά θέματα. με βάση τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από διαφόρους βουλευτές, Προφανώ αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί κάποιε ανησυχίε και ελπίζω ότι θα μπορέσω να σα διευκρινίσω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου και να απαντήσω στις ερωτήσει σα. Η αρχή του κράτου δικαίου και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι βασικέ αρχέ για τη συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες αρχές για τη συνεργασία των κρατών μελών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αρχές ε, είναι και θα παραμείνουν στο μέλλον οι αρχές που θα αποτελέσουν την αφετηρία μας για τη δουλειά που θα κάνουμε στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κατά πολύ και υπάρχουν αρκετές νομικές πράξεις και άλλα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο πρέπει να έχουμε κατά νου τις βασικές αρχές ε, για τη συνεργασία στον τομέα του ασύλου. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που θα προστατεύει τους πολίτες σύμφωνα με την ε, Σύμβαση για τους πρόσφυγες της Γενέβης και σύμφωνα με, άλλους, με άλλες συμβάσεις για την προστασία ατόμων που χρήζουν προστασίας. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις, διάφορες διατάξεις συγγνώμη, που επιτρέπουν την άσκηση των μέτρων αυτών με βάση την αρχή της επικουρικότητας ε, και επίσης δίνει τη δυνατότητα στην, ε, ε, στον επαναπατρισμό ατόμων. Υπάρχουν οι νομικές πράξεις που είναι ο κανονισμός του Δουβλίνου για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουμε το κράτος μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ε, μιας αίτησης ασύλου. Υπάρχει η οδηγία για τις ελάχιστες προϋποθέσεις ε, και κριτήρια και άλλη μια οδηγία που θέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση ετούντων άσυλο και διεθνούς προστασίας και ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη όταν χορηγούν τέτοια προστασία. Αυτές οι νομικές πράξεις θα αναθεωρηθούν και θα ενσωματωθούν σε εθνικό δίκαιο στα κράτη-μέλη και τελικά θα αποτελέσουν ένα συνεκτικό πακέτο. Οι προτινόμενες τροπολογίες θα ακολουθήσουν την οδό της συναπόφασης και αυτή η διαδικασία της συναπόφασης σημαίνει ότι ε, θα έχουν ε, απόλυτη πολιτική βάση μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Για το θέμα της μετανάστευσης θέλω να πω ότι ε, η πρόθεσή μας είναι να επιτρέψουμε την νομότυπη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια μπορούν να επιστρέφουν πάλι κατά νομότυπο τρόπο. Όσον αφορά τα θέματα βασικών δικαιωμάτων, και θεμελιωδών δικαιωμάτων και για, τους, για όσους δεν έχουν το δικαίωμα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι βασικέ αρχέ για όλε τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα συγκεκριμένα να αναφερθώ στου κανόνε που έχουν σχέση με την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος. Αυτό καλύπτεται από την Οδηγία για τις επιστροφέ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2008. Αυτή η οδηγία είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς μια νομοθεσία η οποία θα διασφαλίσει δίκαιες και ανοιχτές διαδικασίες για την επίτευξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών επιστροφής πολιτών από την Ευρώπη. Αυτή είναι μια βασική αρχή και πρέπει να δίνουμε ασφάλεια δικαίου και ανθρώπινη μεταχείριση. Ακόμη, καταβάλλονται προσπάθειες συντονισμού της πολιτικής επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών με την οργάνωση κοινών πτήσεων και οι σχετικές αποφάσεις ξεκίνησαν το 2002. Η χρήση κοινών πτήσεων είναι αποτελεσματικός τρόπος ε, διότι γίνεται αποδοτική χρήση πόρων και θέλω να τονίσω ότι εδώ δεν μιλάμε ε, για συλλογικές αποφάσεις επιστροφής ατόμων. Μιλάμε για συντονισμό δράσεων των κρατών μελών από τη στιγμή που έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις. Η οδηγία που προκύπτει από την απόφαση του Συμβουλίου λέγει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιες πτήσεις για άτομα που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις παραμονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη οργανώνουν την επιστροφή και τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε τέτοιε δράσεις επιστροφής πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε άτομο που επιστρέφει χέρι ε, πλήρους ε, εφαρμογής των δικαιωμάτων του. Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στη Frontex δηλαδή, υπάρχει σχετική οργάνωση για να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη όταν λαμβάνουν μέτρα επιστροφής υπηκών τρίτων χωρών. Τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τη Frontex να εξετάσει εάν μπορεί να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει κοινέ πτήσεις επιστροφής. Ο σκοπός ήταν να διασφαλίσουμε την παροχή διεθνούς προστασίας για αυτούς που χρειάζονται διεθνή προστασία και όταν ε, μιλάμε για επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών, ατόμων που παραμένουν παράνομα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτό θα γίνεται με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τη σωστή νομική διαδικασία. Η οργάνωση κοινών πτήσεων επιστροφής δεν σημαίνει ότι αμφισβητείται η αρχή ε, της μη επαναπροώθησης αναμένεται από τα κράτη-μέλη ότι θα λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές συνθήκες που ισχύουν για κάθε άτομο όταν εξετάζεται η επιστροφή του συγκεκριμένου ατόμου. Και αυτό ισχύει και για άτομα που προέρχονται από το Αφγανιστάν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστροφή είναι πολύ σημαντικέ, αλλά αυτό είναι μία μόνο πτυχή μια ευρύτερη πολιτική μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέρυσι το Σεπτέμβριο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνολική τη προσέγγιση έναντι της μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα θέματα μετανάστευσης πρέπει να θεωρηθούν τμήμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περί εξωτερικών σχέσεων γενικότερα και το θέμα της ε, μετανάστευσης είναι μια συνολική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε καλύτερη εταιρική σχέση με τις χώρες προέλευσης, με τις χώρες ε, διέλευσης και με τις χώρες προορισμού. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο συζητήσαμε σήμερα λίγο πιο πριν, θα επιβεβαιώσει και θα αναπτύξει περαιτέρω αυτή τη συνολική στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Μπιλστρόμ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Μπαρό, εκ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας υπενθυμίσω τις ε, βασικές αρχές που διέπουν την ε, αντιμετώπιση μας για τα προβλήματα αυτά της ε, μετανάστευσης και της επαναπρόθεσης. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν στους υπηκόους ε, τρίτων ε, ε, χωρών μία διεθνή προστασία εφόσον το ζητήσουν. Σε ό,τι φορά τη δυνατότητα οι Αφγανοί αυτοί οι πίκοοι να λάβουν μία ή άλλη μορφή διεθνούς προστασίας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάζουν κάθε αίτηση ασύλου εφαρμόζοντας τα κριτήρια που θεσπίζει η κοινοτική νομοθεσία και λαμβάνοντα υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε αίτηση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν αν ο ετών άσυλο μπορεί να ζητήσει το καθεστώ του πρόσφυγα και αν δεν πληρεί τα κριτήρια που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί ω πρόσφυγα, θα πρέπει να εξακριβώσουν κατά πόσο μπορεί να τύχει τη επικουρική προστασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις αρχές μία προς μία. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να αποπέμπονται στις χώρες τους εφόσον εκτίθενται σε σοβαρές απειλές εκεί. Η κοινοτική νομοθεσία και ιδιαίτερα η οδηγία για το άσυλο προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν την αρχή της μη σε σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Τα κράτη-μέλη δηλαδή δεν μπορούν να αποπέμψουν στο Αφγανιστάν ανθρώπους που είναι πρόσφυγες ε, με τους όρους της συνθήκης της Γενέβης ή έχουν τύχη της επικουρικής ε, προστασίας. Τα κράτη-μέλη άλλωστε ε, υποχρεούνται να βεβαιωθούν ότι καμία τέτοια δράση επιστροφής, επιχείρηση επιστροφής δεν θα γίνει κατά παράβαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τη μη επαναπροώθηση ενός ανθρώπου στη χώρα του αν ε, ε, απειλείται η ζωή του ή η δίωξη εφόσον ε, επιστρέψει εκεί. Επίσης, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα αιτήματα για το κατά πόσο είναι σκόπιμες τέτοιες διαδικασίες απομάκρυσης προς το Αφγανιστάν. Η υπήκοοι του Αφγανιστάν είναι οι τρίτη της χώρας που κατεξοχή ζητούν άσυλο. Και μάλιστα ε, μόνο ένα μικρό κλάσμα τέτοιων αιτήσεων γίνεται δεκτό και οι περισσότεροι βρίσκονται στις γειτονικέ χώρες από το Αφγανιστάν, κυρίως στο Ιράν και στο Πακιστάν. Δεν μπορούμε λοιπόν να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας σε ό,τι αφορά το κατά πόσο η υποχρεωτική επιστροφή Αφγανών στην πατρίδα τους καταστρατηγεί το κοινοτικό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη που δέχονται τις αιτήσει να τις μελετούν διεξοδικά και περιπτωσιολογικά και να αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Κατά την εξέταση των αιτήσεων, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μελετήσουν τις ιδιαίτερες ατομικές περιστάσεις για να κρίνουν κατά πόσο ε, ο συγκεκριμένος ετών ε, έχει ανάγκη επικορικής προστασίας. Φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ανθρωπιστικά, πολιτικά κριτήρια και η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν. Επίσης θα εξεταστεί η ιδιαίτερη κατάσταση του τμήματος της χώρας, περιοχής της χώρας από την οποία κατάγεται ο ετών αλλά και οι ιδιαίτερες ε, δικές του καταστάσεις, η οικογενειακή του κατάσταση, το περιβάλλον, οι δραστηριότητες του στην πατρίδα του ή οποιαδήποτε άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ε, πλέον ευάλωτο. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντλήσουμε κάποια γενικά συμπεράσματα για τις ανάγκες προστασίας των Αφγανών ετούντων. Τα στατιστικά στοιχεία πάντως μας δείχνουν ότι το ποσοστό αναγνώρισης ε, τέτοιων αιτήσεων έχει αυξηθεί το τελευταίο καιρό. Το πρώτο εξάμεινο του 2009 περίπου 70% ε, των Αφγανών ετούντων έχει τυχή διεθνώς προστασίας ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2008 ήταν ε, λιγότερο από 30% ο αριθμός τους. Και θα περάσω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται πριν ε, ληφθεί απόφαση για μια ε, για μια επιχείρηση επαναπρόθεσης. Στην περίπτωση μια κοινή επιχείρηση ε, Μεγάλη Βρετανία Γαλλία ε, στην Καμπούλη, είχα πει ότι πριν επαναπροωθηθεί κάποιο σε μια τρίτη χώρα όπω το Αφγανιστάν, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τρει προφυλάξει. Καταρχήν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο ενδιαφερόμενο δεν, δεν επιθυμεί να τύχει διεθνού προστασία Δεύτερον, αν μια αίτηση διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί, θα πρέπει να βεβαιωθούν τα κράτη-μέλη ότι η αίτηση αυτή όντως εξετάστηκε εις βάθος διεξοδικά και κατά περίπτωση και έχει απορριφθεί μετά από μια κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης. Και τρίτη προφύλαξη, θα πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο η ζωή του μετανάστη αυτή, εφόσον επαναπροθεθεί στην πατρίδα του, δεν ε, θα τεθεί υπό απειλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε διευκρινήσεις για τις περιστάσεις αυτής της ε, κοινή επιχείρησης ε, απομάκρυσης Αφγανών ε, που έγιναν από το, μεγάλο, από Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα στοιχείο που να στοιχειοθετεί παράβαση των τριών αυτών προϋποθέσεων για τους ενδιαφερόμενους. Τι συνέβη λοιπόν αυτές τις διαδικασίες απομάκρυσης ε, για πολύ περισσότερους ανθρώπους. Βέβαια θα, πρέπει η αίτηση, κάθε μια αίτηση να αναλυθεί διεξοδικά. Το πρωτόκολλο 4 της Συνδίκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Θεμελιώδης Χάρτης απαγορεύουν τις συλλογικές αποπομπές, απομακρύνσεις. Αλλά δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα, ούτε καμία, ε, κανένα κόλλημα από τις αρχής ε, ως προς την ε, μεμονωμένη εφαρμογή πολλαπλών μέτρων απομάκρυνσης ε, και την εφαρμογή τους με μια κοινή επιχείρηση. Κάθε όμως ε, τέτοιο μέτρο θα πρέπει να έχει ληφθεί με ξεχωριστή απόφαση ή χρησιμοποιώντας μια κοινή πτήση. Δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για την διεξαγωγή αυτών των επιχειρήσεων από κοινού από διάφορα κράτη-μέλη. Το, η εντολή της Frontex προβλέπει ήδη μια επιχειρησιακή συνεργασία των κρατών μελών στην περίπτωση κοινών επιχειρήσεων απομάκρυνσης. Το Συμβούλιο ζήτησε οι επιχειρησιακές ικανότητες της Frontex να ενισχυθούν και επίσης να ε, ε, υπάρξει δυνατότητα τακτικής συνάβλωσης αεροσκαφών για την διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων. Αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις απομάκρυνσης θα πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τέτοιων δράσεων από άποψη επιμελητίας και να τύχουν και κάποιων συνοδευτικών μέτρων γιατί τέτοιου είδους απομακρύσεις είναι οδυνηρές. Παρόλο που δεν έχει ενσωματωθεί στις κρατικές ένωμες τάξεις η οδηγία για την επιστροφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να βεβαιωθούν ότι οι αποφάσεις τους για την επιστροφή πληρούν τους κανόνες της οδηγίας. Για παράδειγμα, να δίνεται προτεραιότητα στις ε, οικειοθελείς επιστροφές και μάλιστα να προβλέπονται κάποια ένδικα μέσα ή κάποια, κάποιες προσφυγές και να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα πιο ευάλωτων ετούντων. Βέβαια, η οδηγία αυτή δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, αλλά θα εφαρμοστεί όσον οπό και θα επιτρέψει την εφαρμογή περαιτέρω εγγύων υπέρ των ενδιαφερομένων. Αυτές λοιπόν κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ είναι οι απαντήσεις που θα ήθελα να δώσω και που τηρούν φυσικά και επαναλαμβάνουν την κοινοτική νομοθεσία. Όπω είπε και το Μπία Πίλιστρομ, προσπαθούμε για όλα αυτά τα προβλήματα να διασφαλίσουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της ε, επιθυμίας φιλοξενίας και υποδοχής όσων διώκονται για πολιτικούς λόγους και που πραγματικά χρήζουν προστασίας και αξίζουν προστασίας, αλλά να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι ορισμένες αιτήσει είναι α, απαράδεκτες. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ λεπτή ισορροπία και αυτή αναζητούμε ανα πάσα στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά θα ήθελα να σας πω και περιμένω τις απαντήσεις και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ε, Ευχαριστώ κύριε Μπαρό. Τώρα θα δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Δύο λεπτά η κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποδεχθεί τα άτομα τα οποία φεύγουν για λόγους πολέμου ή δίωξης και θα πρέπει να τους εκφράσει, να τους εξασφαλίσει τη διεθνή προστασία με βάση τις αξίες της. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει μεταναστευτικές ροές μεικτέ και υπάρχουν και διακινητές οι, οι οποίοι ε, καταχρώνται τα εθνικά συστήματα και διευκολύνουν την ε, ιζοχή ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στην ε, επικρατειά μας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το θέμα τίθεται στο εσωτερικό κάθε ενός κράτους μέλους. φυσικά το δυναμικό απορρόφησης των κρατών μελών δεν είναι απεριόριστο καθεστώτα προστασίας θα πρέπει να φτιάχνονται για άτομα που πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια. Και αν θέλουμε να κρατήσουμε τις παραδόσεις της χώρας ε, υποδοχής, θα πρέπει να, ε, να εξασφαλιστούμε ότι δεν ε, καταχρώμαστε το σύστημα, δεν καταχρώνεται κάποιοι το σύστημα. Επίσης, χώρες όπως το Αφγανιστάν ή το Ιράκ θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις. Θα πρέπει κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποια και αν είναι η πολιτική τους στάση, να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνένεση, συνένεση ούτως ώστε προσεχώς να υιοθετήσουμε μικτές επιχειρήσεις απομάκρυνσης που θα χρηματοδοτούνται από τη Frontex. Αυτή η πρωτοβουλία ε, είναι ένα κοινό τρόπο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και θα πρέπει να τη χαιρετήσουμε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι ομαδικέ επιχειρήσει απομάκρυνση είναι κάτι διαφορετικό από τι ε, συλλογικέ ε, απελάσει με βάση την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το δικαστήριο του Στρασβούργου ε, απαγορεύει τέτοιου τύπου μέτρα, αλλά τα επιτρέπει όταν τέτοια μέτρα ε, λαμβάνονται μετά από μια αντικειμενική εξέταση της ειδική κατάστασης ε, των ξένων αυτών. Υπηκών. Το Διεθνέ Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για του Πρόσφυγε είναι πυκνό, ούτω ώστε αυτέ οι διαδικασίε απελάσεων να πλησιώνονται σωστά και να γίνονται με το σεβασμό της αξιοπρέπειας και της ακαιρεότητας των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο για δύο λεπτά στην κυρία Σιλβί Γιόμ. Άκουσα πολύ προσεκτικά ε, τους προηγούμενους ομιλητές και θα ήθελα ε, να σας ε, παραθέσω κάποιες ανησυχίες για το θέμα αυτό και θα βασιστώ σε δύο σύντομα πρόσφατα παραδείγματα. Το πρώτο για την απομάκρυνση 27 ατόμων από το Αφγανιστάν προς την Καμπούλ σε μια κοινή επιχείρηση Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας θα ήθελα να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι το Αφγανιστάν είναι μια χώρα όπου η σωματική ακεραιότητα αυτών οι οποίοι ε, απομακρύνθηκαν είναι εγγυημένη η Επιτροπή θα πρέπει να μας πει ότι ε, αυτό έγινε επειδή τα άτομα αυτά δεν είχαν ε, κάνει αίτηση διεθνούς προστασία και κάθε φορά θα πρέπει να μας πει αν ε, έγινε εξέταση των προσωπικών περιστάσεών τους. Δεύτερον, η αποστολή από τη Γερμανία και την Αυστρία ατόμων ε, Ρώμ προς το Κωσυφοπαίδιο ε, παρότι η Διεθνής ε, του ΕΕ για τους πρόσφυγες λέγει από μια πρόσφατη δήλωση παραθέτω ότι, είναι, ότι υπόκεινται η, Ρώμ, η Ρώμα σε απειλές και σε φυσικούς κινδύνους το 4Γ της οδηγίας του 2004 που μιλάει για απειλές ε, κατά ατόμων και για το ε, δικαίωμα σε επικουρική προστασία γιατί το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται ε, στεναρά. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης εάν θεωρείτε επαρκές το να αποστέλλονται, το να επαναπροωθούνται άτομα που δεν έχουν καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας ακόμη και ενώ γνωρίζουμε ότι πολλοί δυνητικοί σε άσυλο δεν κάνουν την αίτηση στην πρώτη είσοδό του, γιατί έχουν πολύ μικρέ πιθανότητε επιτυχία Και άλλη μια ερώτηση, αν τα ε, ε, κράτη-μέλη ε, θα επικυρώσουν την απόφαση του Συμβουλίου τη 29 η 30ης η οκτωβριου σχετικά με τη Frontex και αν τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν για ένα ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών χωρών και αν θα δράσουν για ένα κοινό καθεστώ ασύλου για την εναρμόνιση προς ε, ένα καλύτερο επίπεδο των διατάξεων που έχουν σχέση με το άσυλο και, την, ε, και τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεσάχνε. Ήθελα να μεταφέρω τη θλίψη πολλών Ευρωπαίων γιατί στις 28 Οκτωβρίου δύο ευρωπαϊκές χώρες οργάνωσαν ε, την, επιστροφή, την υποχρεωτική επιστροφή στο Αφγανιστάν 27 Αφγανών και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Ευρώπη πιστεύοντα ότι θα βρουν άσυλο και προστασία. Και του ε, αποπέμψαμε σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την ε, ακαιρεότητά του. Και μάλιστα Ποια ήταν η έκπληξή μου όταν είδα λίγες μέρες μετά ότι, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβλέπει όχι μόνο την οργάνωση κοινών πτήσεων αλλά και τη χρηματοδότησή τους από τον κοινοτικό προπολογισμό, κάτι που αποτελεί καινοτομία. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε κύριε Επίτροπε. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να νομιμοποιεί αθέμητες πρακτικές που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα ο Γάλλος Υπουργό Μετανάστευσης δήλωσε ότι οι υποχρεωτικές επιστροφές θα πρέπει να γίνονται υπό την Ευρωπαϊκή Αιγίδα. Και δεν νομίζω ότι ε, για αυτός ήταν ο σκοπό ε, που είχαν στο μυαλό τους οι πατέρες για την ε, ε, δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, οι Αφγανοί δεν είχαν δυνατότητα να ζητήσουν το άσυλο γιατί οι αιτήσει τους απορρίφθηκαν και μάλιστα ε, η επιχειρηματολογία ήταν ότι η ζωή τους δεν τελούσε υπό απειλή στην περιοχή της καταγωγής τους. Θα ήθελα να μας επιβεβαιώσετε αν έγινε μεμονωμένη εξέταση κάθε αίτηση ατσίλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί το Αφγανιστάν ως ασφαλή χώρα. Γιατί αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο θα ήθελα να μάθω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι αυτή η υποχρεωτική επιστροφή καταστρατηγεί το άρθρο 3 της ε, Σύμβασης της Γενέβης. Και σας ευχαριστώ για τις ε, εξηγήσεις που περιμένω θα δώσετε. Ευχαριστώ. Κυρία μου, θα δώσω εδώ το λόγο στην κυρία Ελέν Φλότρο θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ που γίνεται μια συζήτηση για αυτό το θέμα σήμερα, γιατί είναι σαφέ ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαν προβλέψει ότι η επιστροφή των λαθρομεταναστών που διαβιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Αφγανιστόν ε, θα πρέπει να γίνει ε, με σωστό τρόπο. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Καταρχά, ε, καλό είναι που ζητάμε πληροφορίε από την κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Και χαίρομαι που γίνεται και αυτή η συζήτηση σήμερα για αυτό το θέμα. Τα ερωτήματα έχουν ήδη τεθεί. Το Αφγανιστάν είναι μια ασφαλής χώρα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Ομπάμα, ο οποίο ε, αποφάσισε να στείλει 34.000 στρατιώτε. Κανένα στρατό δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ε, επιβίωση των ε, ανδρών αυτών στο Αφγανιστάν. Θα είμαστε εμεί σε θέση να εξασφαλίσουμε ότι οι μετανάστες που επαναπροωθούμε σε αυτές τις χώρες δεν θα διατρέξουν κανένα κίνδυνο. Αυτό είναι αστείο. Νομίζω ότι και το Γραφείο Προστασίας των Προσφύγων ε, δεν συμφωνεί και σύστησε στα κράτη-μέλη να μην προχωρήσουν σε αυτές τις επαναπροωθήσεις. Κάτι άλλο, για τις μαζικές απελάσεις. Όλοι χαίρονται και εγώ πρώτη για το δεσμευτικό χαρακτήρα της του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, άρθρο 19, 1 και 2. Απαγόρευση αυτών των συλλογικών απελάσεων. Εσείς λέτε ότι δεν είναι συλλογικέ απελάσεις. Ο κ. Μπίλσομ λέει ότι είναι ε, εύλογη κινητοποίηση πόρων. Ε, πρόσφατα, πολύ σύντομα, θα λέμε ότι αυτά τα τσάρτερ ε, κάνουν καλό. Υπάρχουν όρια. Πού είναι αυτά τα όρια. Στο Πάντε Καλέ υπάρχουν πολλοί Αυγανοί και από εκεί ξεκίνησαν και αυτές οι οργανωμένες επιστροφές Αφγανών από τη Γαλλία. Ε, για λόγους επικοινωνιακούς η γαλλική κυβέρνηση αποφασίζει να οργανώσει τέτοιες συλλογικές ε, επιστροφές. Ε, στο πάντο Καλέ της Γαλλίας γίνονται συλλήψεις συλλογικές, παράνομες λοιπόν, γιατί γίνονται διακριτικές μεταχειρήσει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αυτό που λέτε κύριε Μπαρό, ότι πρόκονται για μεικτέ επιχειρήσεις, για άτομα τα οποία ε, δεν βρίσκονται σε νόμιμη κατάσταση μετά από εξέταση ατομικά τη περιπτώσή τους. Όχι, είναι συλλογικές απελάσεις αυτές, ε, μετά από συλλογικέ συλλήψει. Σα ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Κριστίν Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω την οργάνωση αυτής της συζήτησης, όμως λυπούμε για την ξύλινη γλώσσα που ακούγεται, γιατί είναι παιχνίδια λέξεων. Ναι, πρόκειται για συλλογικές απελάσεις. Αυτό οργανώθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Περιφανεύεται ότι τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα ασύλου είναι ένα από αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σήμερα όμως μιλάμε για Αφγανούς οι οποίοι απελάθησαν σε μια χώρα εμπόλεμη, σε ένα πόλεμο στον οποίο συμμετέχουν και πολλέ ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Μπαγό, ζητώ συγγνώμη, αλλά η νομοθεσία περί της οποίας πρόκειται είναι και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εθνική νομοθεσία και μη μας παραπέμπετε στις μεμονωμένες εθνικές περιστάσεις. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών τα οποία συζητάμε έχουν σχέση με τις ε, διατάξεις επιστροφών και αυτή είναι μια οδηγία ντροπή και θέλω να την αποκαλέσω οδηγία ντροπή γιατί είναι οδηγία ντροπή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι το δικαίωμα ασύλου την χάνει διαφορετική μεταχείριση σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και ακριβώς λόγω αυτών των διαφορών οι Αφγανοί δεν είναι σε θέση να ζητήσουν ζητήσουν άσυλο υπό ευνοϊκές συνθήκες. Συμφωνώ λοιπόν με όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι και θέλω να σας ρωτήσω να γίνει αξιολόγηση όλων αυτών των πολιτικών και η δυνατόν ανασυγκεκριμένη πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Στις επόμενες, στις επόμενες παρεμβάσεις με βάση τη διαδικασία Catch the Eye δίνω το λόγο καταρχήν στην κυρία Βεράκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω την κοινή πρωτοβουλία της σοσιαλιστικής βρετανικής κυβέρνησης και της γαλλικής κυβέρνησης που πέπεμψαν και επαναπροώθησαν λαθρομετανάστες Αφγανούς στην πατρίδα τους. Άλλωστε, οι αιτήσει πολιτικού ασύλου που είχαν υποβάλει είχαν απορριφθεί και αυτή η διμερής πρωτοβουλία θα πρέπει να επεκταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί η μεταναστευτική πίεση είναι μια πρόκληση που θα πρέπει συλλογικά να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό το νόημα έχει και το Σύμφωνο Μετανάστευση και Ασύλου που εγκρίθηκε πριν από λίγου μήνε υπό την ε, Γαλλική Προεδρία. Θα πρέπει τώρα να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι ε, αξιοποιώντα τι κοινέ προσπάθειε και ε, χρηματοδοτώντα μέσω τη Frontex κοινέ πτήσει επιστροφών. Και μάλιστα η μελέτη που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πρώτο στάδιο. Θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει αυτέ τι προτάσει, γιατί η καταπολέμηση τη λαθρομετανάστευση ε, είναι προσδοκία των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερα των νόμιμων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι κάθε ετών θα πρέπει να πληρεί διάφορα κριτήρια τα οποία εξετάζονται ατομικά και περιπτωσιολογικά. Όπως ακούσαμε στις προηγούμενες παρεμβάσεις, η εξέταση γίνεται κατά κανόνα με το σωστό τρόπο και όταν οι ενδιαφερόμενοι ε, διαπιστώνουν ότι έχει εξεταστεί ο φάκελός τους, α, Νομίζω ότι παίρνω μια απάντηση. Αυτό που με απασχολεί όμως για το Αφγανιστάν είναι το αν είναι ε, θεμητό να στείλουμε άτομα προς αυτή τη χώρα. Παρά τον ε, ορισμό του ετούντα άσυλο και του πρόσφυγα, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει το δικαίωμα για αυτό το καθεστώς, αν πρέπει να σταλεί προς ε, μια εμπόλεμη χώρα, τότε του δίνουμε το δικαίωμα ε, προσωρινής διαμονής, σε περίπτωση δηλαδή που κινδυνεύει η ζωή του ε, για να, και δεν μπορεί να επιστρέψει εξαιτίας αυτού. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ζέμκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, για τη συζήτηση και να ξεκινήσω από το εξή. Ήμουν εργαζόμουν για πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας και πολλές φορές μετέβη στο Αφγανιστάν γιατί στο Αφγανιστάν υπηρετούν 2.000 Πολωνοί στρατιώτες. Έχουμε λοιπόν ε, εκεί στο Αφγανιστάν ε, ανθρώπους απελπισμένους ε, σε απόγνωση που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και την οικονομική αλλά και την εμπόλεμη. Αλλά και από την άλλη μεριά έχουμε ανθρώπους που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους κυβερνώντες ε, στο Αφγανιστάν και όχι αυτούς που υποστηρίζουν τους Ταλιμπάν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Έχουμε μηχανισμούς και κάποιες ε, δυνατότητες για να αξιολογήσουμε τις ε, πραγματικές προθέσεις και την κατάσταση των Αφγανών που έρχονται στην Ευρώπη. Γιατί ορισμένοι έρχονται από απόγνωση, γιατί βρίσκονται σε διέξοδο, αλλά υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις ε, που τα κίνητρά του ε, δεν είναι τόσο θεμητά. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. είναι περίεργα ορισμένα κομμάτια τη συζήτηση, Γιατί βρίσκονται παράνομα αυτά τα άτομα εδώ. Είναι παράνομα στην Ευρώπη γιατί δεν μπορούν να, βρουν, να βγουν με νόμιμο τρόπο από τη χώρα του που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα δεν είναι αξιοπερίεργο το ότι παρανόμω βρίσκονται εδώ. Και ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανεί αίτηση ασύλου και να ε, γίνει αποδεκτή αίτηση ασύλου. Ε, Ακριβώ ε, διότι η Σύμβαση τη Γενέβη είναι πολύ αυστηρή και πρέπει να αποδείξει κανεί ότι προσωπικά διώκεται. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο όταν φεύγει κανεί από μια εμπόλεμη χώρα Λέμε ότι ε, επειδή δεν έχουν διεκπαιρεώσει την αίτηση ασύλου του πρέπει να τους ξαναστείλουμε στο Αφγανιστάν όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν, να ε, έχουν ε, τα μέσα επιβίωσης και επίσης υπάρχει και πολύ καλό κακό καθεστώς έναντι των γυναικών. Ζητώ λοιπόν από όλα τα κράτη-μέλη και, την Επιτροπή να καταπολεμήσουν αυτές τις επιστροφές προς το Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλείνουμε τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Catch the Eye και θέλω να ζητήσω από τον κύριο Τομπίας Μπίλστρομ να απαντήσει. Herr Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσε παρεμβάσει. σα. Καταρχήν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω κάποιες από τις πιο σημαντικές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό. Ξεκινώ με αυτό που είπε η κυρία Ματιού, όταν μίλησε για αυτές τις μικρές μεταναστευτικές ροές υπάρχουν μεικτές μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εφόσον δεν έχει απεριόριστη δυνατότητα απορρόφησης η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε η κυρία Ματιέ, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την κατά περίπτωση αξιολόγηση για το ποιος χρειάζεται προστασία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις οδηγίες που έχει θεσπίσει έχει και τη γενική εποπτεία αυτών των θεμάτων. Και αυτό έχει σχέση και με αυτό που είπε η κυρία Γκυγιόμ σχετικά με το αν το Αφγανιστάν είναι μια χώρα στην οποία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των ατόμων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται εξατομικευμένη εξέταση κάθε ατόμου και γι' αυτό έχουμε ένα ευρωπαϊκό, ένα κοινό σύστημα ασύλου. Πολλοί ομιλητέ φαίνεται ότι ε, δεν απέδωσαν τη δέουσα σημασία σε αυτό το σημείο. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει το ότι όταν λέμε ναι εννοούμε ναι και όταν λέμε όχι εννοούμε όχι. Επομένως, αν η απάντηση είναι αρνητική, θα πρέπει να διασφαλίζεται και η επιστροφή του ατόμου στην εν λόγω χώρα. Ανεξάρτητα της χώρας για την οποία πρόκειται, θα πρέπει καταρχήν να διασφαλίσουμε ότι το άτομο αυτό είναι ασφαλές και δεν χρειάζεται προστασία και μόνο τότε μπορούμε να αποφασίσουμε με καθαρή συνείδηση ότι θα ξαναστείλουμε κάποιον στη χώρα καταγωγής του. Το αν θα γίνει αργότερα με συλλογικό τρόπο ή αν θα γίνει με μια κοινή πτήση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις που απλώς είναι άτομα που βρίσκονται πάνω στο ίδιο αεροσκάφος. Δηλαδή είναι απλώς θέμα οργάνωσης της πτήσης και δεν είναι συλλογικά μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνονται. Περνώ σε αυτά που είπε η κυρία Κέλλερ, που πάντοτε κάνει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύπλοκο το θέμα, όπως είπατε. Όταν έχουμε ένα σύστημα ε, που λέει ότι πρέπει να βρίσκεται κανείς στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνει αίτηση για άσυλο. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς ε, την αίτηση, είναι δύσκολο να βρεθεί κανείς στην, Ευρωπαϊκή, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποβάλει την αίτηση ασύλου. Και γι' αυτό προωθήσαμε και επί Σουηδικής Προεδρίας ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ούτως ώστε να είναι ε, δυνατόν άτομα τα οποία ενδεχομένως χρειάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό την προστασία, τα άτομα που είναι περισσότερο ευάλωτα δηλαδή, τα άτομα που δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διευκολύνουμε ε, την προστασία τους. Και αν τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να δώσουν ε, όλες ε, ε, τις θέσεις ε, που έχει δώσει η Σουηδία, γιατί εμείς έχουμε διαθέσει 1.900 θέσεις για άτομα που χρειάζονται προστασία. αν μπορούσαν και οι άλλες χώρες να κάνουν τα ίδια εναντί και της είπα της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, νομίζω θα ήταν πολύ αποτελεσματικό. Γιατί έτσι πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Μπαρό. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Η μέγιστη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε προέρχεται από τις μικτές μεταναστευτικές ροές που είπε η κυρία Ματιό. Έχουμε οικονομικού ε, μετανάστε ή μετανάστε που έρχονται για λόγου περιβαλλοντικού και παράλληλα ανθρώπου, οι οποίοι πραγματικά διώκονται και φυσικά έχουν το δικαίωμα σε διεθνή προστασία ή σε ποικρική προστασία. Αυτή είναι η μεταναστε που ερχονται για λογου περιβαλλοντικου Και παραλληλα ανθρωπου οι οποιοι πραγματικα διωκονται και φυσικα εχουν το δικαιωμα σε διεθνη προστασια η σε επικουρικη προστασια αυτη ειναι η δυσκολια και αυτο θα πρέπει να καταλάβουμε για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που θα ήθελα είναι να απαντήσω καταρχήν θα ήθελα να διαβάσω ε, κάποια στοιχεία, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ε, θα ήθελα να διαβάσω κάποια στοιχεία της γαλλικής ε, απάντησης από τη γαλλική κυβέρνηση, γιατί με ρωτήσατε. Διαβάζω λοιπόν τη γαλλική απάντηση. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν είχαν παρουσιάσει αυθόρμητα αίτηση ασύλου ε, και που συλλήφθηκαν σε παράνομη κατάσταση, κρατήθηκαν προσωρινά. Ο καθένας έλαβε στη γλώσσα του μια απάντηση και μπορεί να αντιδράσει στην απόφαση επιστροφής. Ε, και να στραφεί και προς το ε, ε, Γαλλικό Γραφείο Προστασίας των Προσφύγων και των Απάτριδων. Μεταξύ αυτών των ξένων, μόνο ένας δεν έχει απευθυνθεί προς τις γαλλικές αρχές και δύο άλλοι εξετάζονται τώρα οι αιτήσει τους και τους ακούσαμε παρουσία ενός διερμηνέα. Στο διοικητικό δικαστήριο ε, παρουσία διερμηνέα και δικηγόρου παρουσίασαν την περίπτωσή τους και τους κινδύνους που θα, στους οποίους θα εκτίθενται αν επιστρέψουν στην τους, πατρίδα τους. Ε, ορισμένοι Αφγανοί ζήτησαν διεθνή προστασία ή επικουρική προστασία. Ε, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν ότι δεν ε, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρήσουμε ότι θα διωχθούν, ε, ότι αντιμετωπίζει κίνδυνο η ζωή τους σε περίπτωση επιστροφής. Υπάρχει επίσης απάντηση από τη Βρετανική κυβέρνηση. Εγώ έκανα αυτό που απαιτούσε η συνείδησή μου και, το, και η θέση μου. Ζήτησα δηλαδή το λόγο από τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη απάντησαν. Ε, για αυτή την έννοια της ασφαλούς χώρας, τι μπορώ να σας πω. Υπάρχει μια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΔΕΚ που λέει ότι η μόνη περίπτωση που του να προέρχεται κανείς από μια ε, περιοχή ή χώρα που δεν είναι σίγουρη δεν δίνει το δικαίωμα σε διεθνή προστασία ή επικουρική προστασία. Εκτός και αν ο κίνδυνος είναι τόσο υψηλός και υπάρχουν πραγματικές απειλές εναντίον του, του ατόμου, εναντίον της ζωής του. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν από τα εν λόγω άτομα. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω ε, για αυτές τις ομαδικές πτήσεις. Η Frontex οργάνωσε ήδη ομαδικές ε, πτήσεις και χρηματοδότησε εν μέρη αυτές τις πτήσεις. Θα πρέπει να το πούμε. Ε, το 2008 έγινε κάτι τέτοιο, έγινε και το 2009. δεν είναι κάτι το καινοφανέ. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει η Frontex και νομίζω ότι ο διευθυντή της Frontex το κάνει είναι να γίνονται αυτές οι ομαδικές πτήσεις μέσα σε, αξιοπρεπές, σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Να υπάρχει σεβασμός των συγκεκριμένων ανθρώπων. Πρόσφατα μου είπε ο διευθυντής της Frontex ότι παρατήρησε ότι στην Αυστρία υπήρχε ένας διαμεσολαβητής ο οποίος επαγρυπνούσε ούτω ώστε να γίνονται σεβαστές αυτές οι ε, συνθήκες επιστροφής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε. Δηλαδή, να υπάρχει μια εμπειρογνωμοσύνη, μια πραγματογνωμοσύνη, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτά τα οποία επαναπατρίζονται και που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επικουρικούς προστασίας, ε, όταν επιστρέφουν στη χώρα τους να επιστρέφουν ε, μέσα σε σωστές συνθήκες. Αυτό εξετάζουμε, ε, γιατί μας το ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν ε, οργανώνουμε τέτοιε πτήσει χωρί καμία εγγύηση, χωρί σεβασμό των ε, ανθρώπων αυτών. Θα ήθελα να σα πω πάνω απ' όλα το εξή. Ευχαριστώ τον ε, Τομπία Μπίλστρομ και την Σουηδική Προεδρία που μα βοηθάει πολύ. Να σα υπενθυμίσω ότι την Άνοιξη είχαμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε, να φτιάχνουμε το ένα κείμενο που θα μα επιτρέψει να πετύχουμε την Ευρώπη της, του ασύλου. Έχουμε ένα κείμενο για τις συνθήκες υποδοχής, ε, αναφέρθηκε και το Δουβλίνο και πραγματικά θέλουμε να προσαρμόσουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου ούτως ώστε να αποφύγουμε ε, ο κανονισμός αυτός κάποια χρονική στιγμή να χρησιμοποιηθεί εναντίον των συμφερόντων των ευπαθών ατόμων και των παιδιών. Ε, δεχτήκαμε την αρχή κάποιων παρεκκλήσεων στο κανονισμό του Δουβλίνου. Και στις 21 Οκτωβρίου υιοθετήσαμε δύο άλλα κείμενα πολύ σημαντικά το ένα αφορά η Κομισιόν τα υιοθέτησε, έτσι. Το ένα, η οδηγία για τις προϋποθέσεις και την οδηγία για τις διαδικασίες του ασύλου. Και σε αυτά τα σχέδια οδηγιών που είναι καινούρια για το άσυλο, προσπαθούμε να καθορίσουμε κριτήρια τα οποία θα είναι πραγματικά αντικειμενικά, που θα είναι τα ίδια παντού και φυσικά χρειαζόμαστε το Γραφείο Υποστήριξης για να επαληθεύσουμε ότι οι πρακτικές είναι λίγο πολύ οι ίδιε σε όλη την Ευρώπη, ούτω ώστε αυτή η Ευρώπη του ασύλου να αρχίσει να αναδύεται. Ευχαριστώ τη Σουηδική Προεδρία, η οποία νομίζω ότι έχει εισαγάγει στο Συμβούλιο ε, και παρουσιάσει τα διάφορα κείμενα, αλλά τα οποία δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί. Υπάρχουν δυσκολίε. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε να προωθήσουμε την Ευρώπη του ασύλου ε, με τη βοήθεια της Σουηδικής Προεδρίας, η οποία έδωσε και το παράδειγμα ο Τομπίας Μπίλστρομ υπενθύμησε ότι η χώρα του έχει το καθεδρία στην Ευρώπη και έδωσε το παράδειγμα στην Ευρώπη. Γιατί πίσω από αυτό το πρόβλημα υπάρχει μια πιο μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για να υποδεχτούμε αυτούς τους πρόσφυγες και να τους εξασφαλίσουμε την προστασία. Θα πρέπει όλες οι χώρες να βοηθήσουν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν ακόμα χώρες οι οποίες δεν υποδέχονται τέτοια άτομα. Αυτά ήθελα να σας πω έχω συνείδηση και επίγνωση ότι δεν απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Πάντως θα ήθελα να σας πω ότι από πλευράς Κομισιόν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Και ακόμα περισσότερο οι ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. κύριε και κύριοι, μετά την παρέμβαση και του Επιτρόπου, ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Και θα περάσουμε στο επόμενο. Τη δεύτερη